Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθίστε. Ich möchte mit der Sitzung beginnen. Θα ήθελα <clears throat> να μπορέσουμε να αρχίσουμε την συνεδρίαση. Και σε ό,τι αφορά την ημερησία διάταξη, υπάρχουν ορισμένες αλλαγές για αύριο. Θα εκλέξουμε σήμερα έναν ακόμα αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών. Αύριο δε θα δούμε την ύπατη εκπρόσωπο η οποία τα καταφέρνει μετά από την τελευταία φορά που είχε προσέλθει που ήταν η 11η Φεβρουαρίου να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της και να επανέλθει. Ε, και επιτρέψτε μου και εμένα να μην βρω πλέον την δύναμη να την προσκαλέσω ξανά. Ίσως να καταφέρουμε να επιζήσουμε τους δύο μήνες που μένουν και χωρίς την παρουσία της θα σας προτείνω η συμφωνία που αφορά την Ιταλίδα Υπουργό Εξωτερικών που θα παρουσιάσει αύριο την Ιταλική Προεδρία να παραμείνει και να μας εξηγήσει και τα σχετικά με το άτυπο Συμβούλιο Γκίμνιχ. Θα έρθει ήδη από τις 9. 9 αύριο λοιπόν το πρωί αρχίζει η συζήτηση με την κυρία Μοργκερίνη. Ε, θα καταφέρω να προφέρω και το όνομά της κάποια στιγμή σωστά. Μέχρι τις 10.30-11 περίπου θα ακολουθήσουν οι συνομιλίες με τα άλλα πρόσωπα που προβλέπονται στην ημερησία διάταξη. Με τον ε, πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ. Για την Ουκρανία θα μιλήσουμε με τον κύριο Αρμπακάν που είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΟΑΣΕ και τον κύριο, και τον κύριο Πίτερ Μπάλας της ομάδας στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά θα έχουμε και τα θέματα του προϋπολογισμού. Αν συμφωνείτε λοιπόν με την ημερησία διάταξη ως έχει, τότε νομίζω μπορούμε να την εγκρίνουμε. Αν δεν προβάλλεται καμιά ένσταση τότε εγκρίνεται η ημερησία διάταξη και έχω να ανακοινώσω ακόμη ότι και στις θερινές διακοπές δεν μείναμε άπρακτοι. Ο πρόεδρός σας έκανε πολλά ταξίδια από το Κίεβο μέχρι την Ράμαλα, μέχρι την Ιερουσαλήμ και συνεδριάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέσα του μηνός, του μηνός Αυγούστου κάναμε τηλεφωνική διάσκεψη με προέδρους άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών για να συζητήσουμε τα σχετικά θέματα και την περασμένη πέμπτη για την προετοιμασία του ατύπου Συμβουλίου Γκίμνιχ όπου μπόρεσα να συμμετάσχω εν μέρη για να συζητήσουμε με το Συμβούλιο για θέματα Ιράκ-Συρίας από τη μια μεριά και Ουκρανίας από την άλλη. συμμετέσχει και εκπρόσωπος του Διευρυμένου Προεδρείου της παρούσας Επιτροπής Εξωτερικών, αλλά και εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών επιτροπών που ανέφερα προηγουμένως. Θα συνεχιστεί η συζήτηση αυτή και σήμερα και αύριο διότι είναι αρκετά δραματική η κατάσταση, όσοι γνωρίζετε, και στην μακρά ενεργό πολιτική μου ζωή, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχω ξαναζήσει τέτοιες δραματικές καταστάσεις. Τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία σημαίνουν απλά ότι σε ευρωπαϊκό έδαφος διεξάγεται πάλι πόλεμος. Γίνεται εισβολή ξένων δυνάμεων σε άλλη χώρα. Κάποιοι προσπάθησαν να πούν ότι πρόκειται για κάποιους αδιούχους στρατιώτες οι οποίοι έκαναν λάθος και πήραν λάθος δρόμο και μπήκαν με τα τάγκς στην Ουκρανία. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Γίνεται πραγματικός πόλεμος. Θα το συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε ακόμη και τα όσα έχουν σχέση με τις κυρώσεις. Ακούω ειδήσει από διάφορες πρωτεύουσες και αυτό το βρισκό δυνηρό. Από την προηγούμενη εβδομάδα ζούμε μια αλλαγή στην Ευρώπη. Βλέπουμε να ξαναπέφτει το σιδηρούν παραπέτασμα. Το ερώτημα που τίθεται είναι πού ακριβώς. θα έχουμε και την σημαντικότερη διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ των τελευταίων 20 ετών, την Πέμπτη. η διασφάλιση της ειρήνης και της ελευθερίας των ευρωπαϊκών λαών πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από μας. Και δεν πρέπει να λογαριάσουμε ποια χώρα ενδεχομένως θα λάβει μεγαλύτερη ζημιά από τις κυρώσεις προς την Ρωσία από τις άλλες. Ο Πούτιν παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τη συζήτηση αυτή. Και τέτοιου είδους διαφωνίες του δείχνουν ότι μπορεί να συνεχίσει όπως έκανε με την Κρυμαία, παρά τις κυρώσεις, όπως έκανε, κάνει τώρα με την Ουκρανία. Τώρα συνεχίζονται οι κυρώσεις βαθμιδών, ο ίδιος συνεχίζει να γρά, όπως θέλει, δεν ξέρω πού θα λήξει το νήμα αυτό. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αυτά τα συνηθισμένα παιχνίδια ιδεών που κάνουμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να συνεχιστούν. Για μένα πάντως το όραμα της διαρκούς ειρήνης που είχα από το 89-90 για την Ευρώπη έχει λήξει. Και οφείλω να ομολογήσω ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα είχα λάθος εκτιμήσει την κατάσταση. Πιστεύω δεν θα πρέπει να πούμε αν ήταν σωστό ή όχι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Καμιά φορά τα πράγματα έρχονται διαφορετικά από ό,τι τα φαντάζεται κανείς. Και αυτό οφείλουμε να το λάβουμε υπόψη. Και όσο ταχύτερα το λάβουμε υπόψη, το, τόσο ταχύτερα θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, που εγκρίνεται το σχέδιο ημερησίας διατάξεως και τώρα για τα πρακτικά αν δεν υπάρχουν στάσεις εγκρίνονται και αυτά. Έχουμε στην εκλογή του Δευτέρου Αντιπροέδρου. Η ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς έχει ανακοινώσει το όνομα του κυρίου Χαβιέ Κούζο, την, ο οποίος θα αντικαταστήσει την κυρία Μαρίνα Αλβιόλ. Ναι, προτείνουμε τον Χαβιέ Ζωπερμούρη, ο οποίο γεννήθηκε στο Φερόλ της Γαλλικής στην Ισπανία. Από το 1980 διαδραμάτισε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο κίνημα κατά του φασισμού και του ρατσισμού ε, για την διεθνή ελληνική και έχει δώσει αγώνα ε, για να μείνουν ατιμόρυτοι εγκληματίες πολέμου. Ανθρώπινα δικαιώματα, γεωπολιτική, και ζητήματα άμυνα έχει ασχοληθεί με αυτά. Επίση, από επαγγελματική έχει πρόσφατα δημοσιεύσει ε, ένα βιβλίο για την νότιο Αμερική και τι ε, αλλαγέ που γίνονται εκεί. Οπότε, ο κύριο Κούσο επίσης εργάζεται στην Υποπιτροπή για άμυνα και ασφάλεια, στην αντιπροσωπεία για τη σχέση με το Ιράκ και με την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Ε, Προκαλώ να επιβεβαιωθεί η πρώτη ως αντιπρόεδρος για τη δική μας παράταξη. Σας ευχαριστώ κυρία συνάδελφε. Δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα. Ζητεί κανείς να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία. Δεν έχει μικρόφωνο ο κύριος βουλευτής. Δεν έχει μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, ο και κ. Μπεσίρ πρόκειται να λάβει τη θέση του αναπληρωτή στη θέση της κυρίας Κουκούλη. Το σημειώνουμε, ευχαριστώ. Κύριε Τάνοκ. Εμείς δεν έχουμε λάβει γνώση αυτών των μεταφορών για το Προεδρείο. Είναι κάτι ε, το οποίο γνωστοποιήθηκε. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τι έγινε δεν είναι, τι έγινε, σαν να μην ήμασταν ε, εδώ το καλοκαίρι, σαν να ήμασταν βουλευτές το καλοκαίρι. Εάν έχω κατανοήσει καλά, ήδη είχε ανακοινωθεί από την τελευταία περίοδο συνόδου της Ολομέλειας από την ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς. Άρα πρόκειται για συνήθη διαδικασία, εάν δεν ζητεί κανείς να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία, τότε προτείνω να ψηφιστεί, να εκλεχθεί ο συνάδελφος δια βοής. Συγχαρητήρια κύριε Κούζο, παρακαλώ προσέλθετε να εγκατασταθείτε εδώ. Äh, sorry. Äh, συγγνώμη, επειδή λόγω της ακροάσεως δεν έχουμε καθίσματα ελεύθερα μετά την ακροάση. Είδα τους μελλοντικού πρέσβεις να ταράσσονται διότι θα χάσουν τις θέσεις τους. Το υπαριθμόν 5 τώρα. Ο πρέσβης κ. Σβάισγκουτ που μέχρι τώρα εκπροσωπούσε τα συμφέροντα της Ένωσης στην Ιαπωνία, και τώρα διορίζεται επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ενώσης στην Κίνα και τη Μογγολία. Για την σημασία του χαρτοφυλακίου αυτού, σε ό,τι αφορά θέματα εξωτερικής πολιτικής και εμπορίου, φυσικά δεν χρειάζεται να επεκταθώ ιδιαίτερα. Ο κ. Κούτ ήδη έχει παρουσιαστεί εδώ ενώπιον μας και είχε παρουσιάσει τα πεπραγμένα του τότε ως πρέσβη στην Ιαπωνία. Θα δούμε τώρα εάν διατηρεί τις ικανότητές του. Κύριε Σφαρισκούτ, χαίρομαι που